συναφές θέμα των Συρίων προσφύγων που έρχονται στα σύνορα της Βουλγαρίας. Και ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Βενιζέλος, εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζει η Βουλγαρία, όπως φυσικά και οι άλλες χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ιδίως στην νοτιοανατολική ευρώπη συνδέονται στενά με την επιδείνωση της κατάστασης στη συρία. λόγω της γεωγραφικής της θέσης η βουλγαρία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. είναι ένα από τα κράτη μέλη που είναι εκτεθειμένα ιδιαιτέρως στις συνέπειες της συριακής κρίσης. το συμβούλιο έχει λάβει γνώση της πρόσφατης έκθεσης του ιανουαρίου του 2014 της ΥΠΑ της αρμοστίας του οργανισμού ηνωμένων εθνών για τους πρόσφυγες. η έκθεση αυτή αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα τα οποία χρειάζονται διεθνή προστασία και αυτό συνδέεται φυσικά και με τη βουλγαρία ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται τα άτομα αυτά. παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί και από ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περιτεύει να υπογραμμίσω ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι οι συνθήκες υποδοχής συνάδουν με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. αναγνωρίζουμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που δέχονται πρωτοφανή ροή ατόμων υπό τέτοιο καθεστώς. οι βουλγαρικές αρχές ιδίω έχουν δηλώσει στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο την προθυμία τους να ανταποκριθούν καταλήλως και επαρκώς. εν οι εγκαταστάσεις υποδοχής είναι περιορισμένες είναι ήδη υπερπλήρης, η ανταπόκριση συνεπώς στις ανάγκες των ατόμων που προέρχονται από τη συρία αποτελεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη πρόκληση. η έκθεση της ΥΠΑ της αρμοστίας του οηε στην οποία αναφέρομαι τονίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί για να προσδιοριστούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας επιπλέον ατόμων που χρήζουν προστασίας καθώς και για να καθοριστούν οι τρόποι που θα καταστήσουν λειτουργικές τις εγκαταστάσεις αυτές. επίσης η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. η επιτροπή όπως φαντάζομαι θα πει η ίδια οργάνωσε αποστολή στη βουλγαρία την προηγούμενη εβδομάδα για να εκτιμήσει την κατάσταση εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα είναι σε θέση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαπιστώσεις της. εκτιμούμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και την ανησυχία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. γνωρίζω ότι ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου επισκέφθηκαν σχετικά πρόσφατα τη βουλγαρία προκειμένου να διαπιστώσουν τις προκλήσεις που η χώρα αυτή αντιμετωπίζει. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στα σημεία εισόδου στην ευρωπαϊκή ένωση των ατόμων που εγκαταλείπουν τη συρία. γνωρίζουμε ότι υπάρχει αριθμός πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί στον τομέα αυτό και ότι η συμβολή τους όσον αφορά τι εγκαταστάσει διάσωση και βοήθεια είναι πολύτιμη. η ευρωπαϊκή ένωση παρέχει επίση πρακτική βοήθεια στη βουλγαρία. 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά έχουν διατεθεί για τη συνδρομή στα κράτη μέλη που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στι μεταναστευτικέ πιέσει και ροέ προκειμένου να βελτιώσουν τι εθνικέ του δυνατότητε. αυτή η χρηματοδότηση περιορισμένη βέβαια έχει ω στόχο τη βελτίωση τη δυνατότητα υποδοχή, τη δυνατότητα διαχείριση, τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφή καθώ και τη υποστήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συνόρων. το συμβούλιο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία που απαιτείται για την ανακούφιση του πόνου των σύριων πολιτών που αναζητούν προστασία και υποστήριξη εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. η βουλγαρία είναι ένα από τα περισσότερο εκτεθειμένα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης σε αυτές τις πιέσεις και ως εκ τούτου είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κάθε μέτρο που θα μπορούσε να συνδράμει τις βουλγαρικές αρχές στην αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων και να τις βοηθήσει στην προσπάθειά τους να παράσχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα που χρήζουν προστασίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. σας ευχαριστώ, η Επίτροπος Μάλστρομ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Η Κομισιόν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές πιέσεις στα συνοριακά κράτη της Ένωσης, κυρίως στη Βουλγαρία. Πρέπει να τονίσω τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η βουλγαρική κυβέρνηση στη συνεργασία με την Κομισιόν, την ΕΑΖΟ, την, τον ΟΙΕ και άλλα κράτη-μέλη, ώστε να αποφευθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, η οποία έχει κάπως οριοθετηθεί, έχει σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον δεν επιδεινώνεται. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές σοβαρές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, η κατάσταση των μεταναστών και των ετών των άσυλο στα καταλήματα. υπάρχει ε, μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την ε, ε, επεξεργασία των αιτήσεων και των όσων έχουν ήδη διεθνές καθεστώς και έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη Βουλγαρία βάλωτος ε, χαρακτήρας των ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία αλλά και η δυνητική, ε, ο δυνητικός αντίκτυπος στη σωστή λειτουργία του κανονισμού του Δουβλίνου είναι προφανές πως η κατάσταση στη Βουλγαρία χρειάζεται επίγουσα δράση. Μπορεί να είναι η πρώτη ευκαιρία για να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό κρίσης, διαχείρισης κρίσης, το άρθρο 23 του κανονισμού Δουβλίνου 3. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίζεται από το άρθρο 23 δεν έχει το νόημα του να κατηγορήσει οποιαδήποτε χώρα και αυτό το, ε, το δικό σας σώμα το γνωρίζει αυτό πολύ καλά ως νομοθέτης. Είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης. Για ενεργοποίησή του θα αναγνώριζε την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης πίεσης σε κάποια χώρα, προσφέρει πολιτική και υλική λύση για το εθνικό σύστημα που πιέζεται αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες, τους ετούντε άσυλο. Το, η χρήση του άρθρου 33 θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα πως η Βουλγαρία δεν είναι μόνη και ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη είναι δεσμευμένα να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να ξεπεράσει την κρίση. Είναι μια έκκληση ε, για αλληλεγγύη με τη Βουλγαρία που μπορεί να πάρει πολλές μορφές, υλική, ε, επιχειρησιακή αλλά και οικονομική συμβολή. Όσον ε, εφόσον έχουμε ήδη υποστήριξει τη Βουλγαρία φυσικά ως Ένωση και μια τέτοια απόφαση πρακτικά θα σημάνει ότι η Βουλγαρία σε συνεργασία με την Κομασιόν και την ΙΑΖΟ θα αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης σε σχέση με τις ανάγκες και τα θεμέλια του πλάνου δράσης ήδη υπάρχουν. Δεδομένων των ε, εμπλεκομένων φορέων, IOM, ΑΖΟ, Κομισιόν, ΜΚΟ, διάφορα κρατημέλη αλλά και τρίτες χώρες, το πρόγραμμα δράσης παρέχει ένα μέσο ώστε να, ε, να, να διαχειριστούμε τα διάφορα μέσα για να αποφύγουμε διαρθρωτικά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος του Δουβλίνου. Επίσης το πρόγραμμα δράση θα εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη ε, πολιτική στο, και την ένταξη των ε, ετών των άσυλο για όσους μείνουν στη Βουλγαρία και θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν νέες κρίσεις στο μέλλον. Η ανάγκη για μακρόπνο προγραμματισμό είναι φυσικά προφανής. Τέλος, ένα τέτοιο πλάνο θα επέτρεπε περαιτέρω επίγουσα βοήθεια αν αυτή είναι απαραίτητη και θα πρέπει να καλύπτει τόσο την άμεση φάση ανταπόκρισης ενώ η στήριξη συνεχίζεται και ε, για την περίοδο μετά από τώρα και φυσικά η Κομισιόν θα συνεχίσει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βέμπερ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Τις τελευταίες ε, ημέρες συζητάμε την κατάσταση στη ε, Συρία, την τραγωδία ε, στην Συρία. Όμω με τη σημερινή ημέρα και τη σημερινή συζήτηση το θέμα μετατίθεται στην Ευρώπη, γιατί μα χτυπάνε την πόρτα άνθρωποι και μα βοηθούν, για να, και μα δουν βοήθεια. Σε ό,τι αφορά του πρόσφυγε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση, γιατί αυτό θέτει την ανθρωπιά της Ευρώπης και την ανθρωπιστική βοήθεια σε δοκιμασία. Την τελευταία εβδομάδα διαβάσαμε στι εφημερίδες άρθρα ε, για την ε, Βουλγαρία, για τους, το, το τείχος, για τις φράχτες που ε, υποτίθεται ότι πρέπει να αποκρούσουν τους πρόσφυγες από τη Σωρία. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Αυτή η εντύπωση που δίδεται ότι οι Ευρωπαίοι κλείνονται σε τείχος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό θέλουμε λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Βουλγαρία έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη γιατί είναι στα σύνορα με τις περιοχές αυτές της κρίσης και ζητώ, κάνω έκκληση στην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Βουλγαρίας για να μην χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό για εσωπολιτικά ζητήματα. Ελπίζω οι πολιτικές ισορροπίες να μην οδηγήσουν στη χώρα στο να μην βοηθηθούν τελικά οι πρόσφυγες από τη Συρία. Η στάση του ΕΛΚ είναι σαφής. Πρόκειται για πρόσφυγες που αξίζουν ε, την υποστήριξή μας. Ε, ζητούμε και από την Τουρκία να συνεργαστεί για την επίλυση των προβλημάτων. Θέλουμε να τηρηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως είπε και η Επίτροπος. Και ε, πρόκειται να δεσμευτούμε για οικονομική αλληλεγγύη με τα κράτη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούμε και στις από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν τη, τον όγκο των ε, προσφύγων από τη Συρία για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Θα πρέπει να δράσει από κοινού η πρόσφυγη. κύριε Βέμπερ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Κύριλοφ θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Κύριος Κύριλοφ, έχει το λόγο. Κύριε Βέμπερ, ως ε, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος σας συνεχίζετε να αναφέρετε ε, τα ίδια πράγματα. Όμως ε, το 2011 είχε προβλεφθεί ε, ο έλεγχος και η υλοποίηση ενός στρατοπέδου για χίλιους ανθρώπους. Όμως είναι δύσκολο να πει κανείς ποια είναι τα μέσα τα οποία απορροφήθηκαν διότι διαπιστώσαμε πως δεν είχε γίνει τίποτα εδώ μεταξύ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει θαύματα μέσα σε λίγους μήνες για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και θα ήθελα να πω ότι η Βουλγαρία όντως από την Βουλγαρία στα εξωτερικά της σύνορα ζητούνται πάρα πολλά αλλά η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει για, στο ερώτημα του γιατί τίθεται το θέμα αυτό, γιατί δημοσιεύονται αυτά τα άθρα, γιατί υψώνεται αυτός ο τείχος και το, τα ακροδεξιά κόμματα όπως το κόμμα ΤΑΚΑ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω και οι σοσιαλιστές εδώ να ασκήσουν επαρκή κριτική στην κυβέρνησή τους. Αυτό ζητούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Γκίγιομ. Σα ευχαριστώ. Πριν από δύο εβδομάδε με διάφορου συναδέλφου. Ε, μεταβήκαμε σε μια αποστολή στη Βουλγαρία μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, της οποίας στόχοι ήταν πολλαπλή, αλλά ανάμεσα σε αυτού ήταν να αξιολογήσουμε επιτόπου την κατάσταση των ετών των άσυλων, να εκτιμήσουμε τι βελτιώσει τη υποδοχή και να προτείνουμε, αν είναι αυτό απαραίτητο, βελτιώσεις ε, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, είναι μοιρασμένε οι εντυπώσεις μας. Από τη μια πλευρά, σίγουρα οι βουλγαρικές αρχές έχουν καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσουν την κατάσταση υποδοχής, Όμω θα πρέπει να διαπιστώσουμε δυστυχώ ότι η κατάσταση επιτόπου, αν και διαφέρει από την αρχή εκεί, εξακολουθεί να είναι δύσκολη και πόρο απέχουμε από αποδεκτή κατάσταση σε ανθρώπινο επίπεδο ή ακόμα και από τα επίσημα στάνταρ για τα δικαιώματα των προσφύγων. Έχω λοιπόν διάφορε παρατηρήσει να κάνω σε σχέση με τι δυσκολίε που διαπιστώσαμε επί το ΑΠΟΥ. Καταρχήν, η πρώτη παρατήρηση αφορά το μηχανισμό για τον οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, κυρία Επίτροπε. Αν ο αριθμό των ετούντων άσυλο που ολοπλασιάστηκε επί 8 σε σχέση με το προηγούμενο έτη, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο το επίπεδο της ζήτησης που είναι προβληματικό, αλλά και η φύση του βουλγαρικού συστήματος που δεν ήταν εξοπλισμένο για να αντέξει μια τέτοια αύξηση αιτήσεων, ε, τόσο όσον αφορά την υποδοχή, όσον αφορά και την διαδικασία. Και καταλαβαίνω ότι μιλήσατε για την ε, ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπει έναν μηχανισμό, αλλά η κατάσταση πιστεύω είναι κατάλληλη. Από τις αρχές του 2013 πολύ ε, αυξήθηκαν οι μετανάστες, η, τάση αυτή έχει ανατραπεί από τον Νοέμβριο και μετά. Η Κομισιόν συνεργάζεται με τις βουλγαρικές αρχές ώστε να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία θα, έχουν, θα, ενταχθούν όντως στη διαδικασία ασύλου και δεν ε, διώχνονται. Και τελευταία μου παρατήρηση. Είναι προφανές ότι η Βουλγαρία ε, πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και, σε και τα θέματα ασύλου. Αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί και η ελληνική τη υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά την υποδοχή των Σύριων προσφύγων με οικονομικό αλλά και με πραγματικό, πραγματική υποδοχή των ανθρώπων. Sorry, ναι, συγγνώμη. Ένα... Στάνει μία, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε μία μπλε κάρτα. Έτοιμα για μπλε κάρτα. Κύριε Στάλινοφ, συνεχίστε παρακαλώ. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να μην συλλαμβάνονται οι πρόσφυγες που επιτρέπει η Τουρκία να περάσουν στη Βουλγαρία. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα αναλάβει εκ μέρους του σοσιαλιστή Προέδρου της Γαλλίας ποιος θα αναλάβει το βάρος να υποδεχτεί ε, άτομα από τη Βουλγαρία και πόσους γιατί προφανώς η Βουλγαρία δεν μπορεί να τους υποδεχθεί όλους να σας πω πως είναι πρόεδρος της Γαλλίας και όχι σοσιαλιστής πρόεδρος ο πρόεδρος μας, είπε πόσους Σύριους μπορεί να υποδεχτεί η χώρα μας. Και μάλιστα θα ξεκινήσει σύντομα. Το θέμα εδώ θα πρέπει ε, να είναι πως τα άτομα αυτά τα οποία παρουσιάζονται στα σύνολα δεν θα επαναπροωθούνται προς τα πίσω από τη στιγμή που όντως χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ευχαριστώ κύριε Σίλτσεφ τώρα.

Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως εγώ πήγα σε δύο αποστολές και στην ε, Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία έχω επισκεφθεί αυτές τις εγκαταστάσεις και η χώρα μας κάνει μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων μας. Αυτοί οι μετανάστες όντως χρήζουν ε, ε διεθνούς προστασίας και θα πρέπει να τους προσφέρουμε καλές συνθήκες ζωής και όχι μόνο στη χώρα της Βουλγαρίας αλλά και, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Βουλγαρία η οποία θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του σε θέματα ασύλου, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα σύνορά μας εκτός από τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Έχουμε τους υπηκόους της Βουλγαρίας οι οποίοι δεν αντέχουν ε, το βάρος αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα και οδηγούμε στο εξή ερώτημα. Πώ θα προστατεύσουμε τα βουλγαρικά σύνορα έτσι ώστε η χώρα μα να προστατευτεί από την είσοδο εγκληματιών, για παράδειγμα. Δεύτερον, πώ μπορούμε παρόλα αυτά να βοηθήσουμε όσου προσπαθούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη που λέγεται Συρία. Η Βουλγαρία αναγνωρίζει τις ανθρωπιστικές τους ανάγκες και ξέρει πως πρέπει να δείξει αλληλεγγύη. Εμείς όμως χρειαζόμαστε τα οικονομικά μέσα που θα μας το επιτρέψουν. Δεν έχουμε τα χρήματα για να τους βοηθήσουμε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Η βουλγαρική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τα κονδύλια του εθνικού προπολογισμού, αλλά χρειαζόμαστε μη κάποιο είδους πολιτική ευελιξία εκτός από τα χρήματα που είναι απαραίτητα. Ζητήσαμε από την Τουρκία να κάνει αυστηρωτά του ελέγχου στα άτομα τα οποία περνάνε μέσω των ε, τουρκικών εδαφών προς τα ε, τουρκικά-βουλγαρικά σύνορα. Αυτή τη στιγμή Έχουμε χιλιάδε πρόσφυγε που καταφθάνουν στα σύνορά μα και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να μα δείξετε αλληλεγγύη για να μπορέσουμε και εμεί να δείξουμε αλληλεγγύη. Και πιστεύω πω το θέμα αυτό θα πρέπει να λυθεί με κάποιο λογικό τρόπο, έτσι ώστε να καταφέρουμε τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό να του ενσωματώσουμε. Γι' αυτό η Βουλγαρία ήδη έχει ξεκινήσει με ένα εθνικό σχέδιο. Ε, ένταξης. Και επαναλαμβάνω υπάρχουν και οι βάσιμες ανησυχίες των ε, πολιτών μας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα. Αυτό που πρέπει να στείλουμε ως μήνυμα είναι πως δεν είναι μόνο η Βουλγαρία στη μάχη αυτή. Μπλε κάρτα από την κυρία Έρνστ. Έχετε το λόγο και 30 δευτερόλεπτα. Έχω μπερδευτεί λίγο, κύριε συνάδελφε, και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλητριάς. Ήθελα να ρωτήσω ποιον εννοείται. Μιλάτε για Σύρους ε, πρόσφυγες ή για άλλα άτομα τα οποία βρίσκονται στα σύνορα, για παράδειγμα, στην... και θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιους αναφέρεστε, δεν έχω καταλάβει. Το 80% των ανθρώπων που βρίσκονται στην Βουλγαρία θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Γιατί η Βουλγαρία είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο όραμα ή αν έχουν πέσει θύματα προπαγάνδας. Παντούς το 80% των ε, προσφύγων μας λένε θέλουμε το καθεστώς του πρόσφυγα να μας χορηγηθεί για να μπορέσουμε να φύγουμε στην Ευρώπη. Αλλά δεν χρειαζόμαστε πια τύχη, ε, δεν χρειαζόμαστε πια ε, φράχτες. έχουμε αυτά τα χιλιόμετρα φράχτη που δεν επιτρέπει στους πρόσφυγες να περάσουν στη χώρα μας. Γιατί, Γιατί οι μετανάστες αυτές, οι μετανάστες, μετανάστες πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να περάσουν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε ε, Βενιζέλ, ε, κυρία Μάλστομς, είναι προφανές πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη πρέπει να βρουν μια καλύτερη λύση για, την, για το Συριακό, αλλά και για να μπορέσουν να ανακαλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων και των ετούντων άσυλο εδώ στην Ευρώπη. Παρατείνεται αυτή η διαδικασία, αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και θα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο και μετά να τους εγκαταστήσουμε. Δεν δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό στην αρχή, αλλά θα είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να τακτοποιήσουμε τους πρόσφυγες ε, με τάξη. Τα κράτη-μέλη ανέκαθεν ε, θέλησαν να αρνηθούν τη βασική αρχή της αλληλεγγύης για τους, για τους πρόσφυγες, αλλά και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και σύμφωνα με τις εκκλήσεις της Επιτρόπου ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου, γιατί δεν πρόκειται μόνο για αλληλεγγύη για το, προς τους πρόσφυγες, αλλά προς ένα κράτος μέλος, τη Βουλγαρία, που αντιμετωπίζει κρίση, όπως και η Ελλάδα. Και ο Υπουργός Βενιζέλος το ξέρει πάρα πολύ καλά το τι έχει περάσει η Ελλάδα. Ε, άρα λοιπόν και το άρθρο 80 των συνθήκων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτές τις περιπτώσεις, όμως το Συμβούλιο ποτέ δεν θέλησε και είπε ότι το 80 που ορίζει την αλληλεγγύη των κρατομελών ήταν προγραμματισμένο και ότι χρησιμοποιούταν πάντα. Αν δεν χρησιμοποιούταν πάντα, θα πρέπει όμως τώρα πλέον να χρησιμοποιηθεί για στρατηγικούς ε, λόγους, για λόγους αρχής, αλλά κυρίως για ανθρωπιστικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δεχτούμε τους πρόσφυγες, ε, να ξεκινάμε από, ήδη από τα σύνορα της Συρίας και να έχουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση για να μην συνεχίζεται ε, άλλη μια τραγωδία μετά την τραγωδία της Συρίας μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία, Ένιστο. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ τι θα πρέπει ακόμα να συμβεί για να καταλάβουμε ότι η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε μία ημέρα ακόμα. Προφανώς ε. η αντιμετώπιση των προσφύγων από τη Συρία στη Βουλγαρία είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και άλλο ένας φράχτης, άλλο ένα τείχος είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Αλλά σας ε, ρωτώ με ειλικρινία. Σχέδια δράσης, πολιτική Τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το άσυλο, τα πακέτα, όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει τίποτα στην, στάση, στην κατάσταση των προσφύγων. Δεν έχουμε προχωρήσει προς μια πιο ανθρώπινη πολιτική. Το Δουβλίνο 3 είναι ένα συνώνυμο για μια πολιτική που δεν σέβεται τον άνθρωπο. Ε, και μιλάμε για την Βουλγαρία, θα μιλήσουμε σε μία ώρα για την Ελλάδα. Μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε και να διαπιστώσουμε μεγάλα ελλείμματα. Και βλέπουμε όταν ε, στο Κοινοβούλιο αποφασίσαμε περικόπη των δαπανών του προπολογισμού, περικόπηκαν και οι δαπάνε για το άσυλο. Για να ξεφορτωθούμε τους πρόσφυγες. Ε. Αυτή την ε, κατάσταση την έχω βαρεθεί πια. Να μιλάμε, να μιλάμε και να μην αλλάζει τίποτα τελικά για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Στογιανό. Κύριε Πρόεδρε, Η ώρα που έχει προβλεφθεί για αυτή τη συζήτηση είναι σκανδαλωδώς ε, σύντομη. Είπατε κύριε Επίτροπη βοήθεια για την ένταξη και την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων που επιθυμούν να μείνουν. Μα πρόκειται για πρόσφυγες που μένουν ε, στην επικράτεια της Βουλγαρίας διότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο ε, στη χώρα τους. Όταν ο κίνδυνος αυτός θα πάψει να υφίσταται θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Για ποια ένταξη λοιπόν μιλάμε. Έπειτα, απάντηση στην ερώτησή μου. Άκουσα, περίμενα μάλλον τρεις φορές για την απάντηση και είπα, υπόθηκε πως η Βουλγαρία είχε δώσει 300.000 ευρώ για να βοηθήσει τις ε, χώρες γύρω από τη Συρία, τις ε, γειτονικές χώρες. Όμως η Βουλγαρία τι πήρε σε αντάλλαγμα. Και να επαναλάβω άλλη ε, μια φορά την ερώτηση. Θα δείξετε πως η Βουλγαρία δεν είναι μόνη της σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί μέχρι στιγμής το αντίθετο έχετε κάνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να καθησυχάσω τον κύριο Στογιανόφ εξ αρχής ότι στην αποστολή αυτού του κοινοβουλίου που μας ε, οδήγησε στη Βουλγαρία πριν από λίγες εβδομάδες, το πρώτο που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ήταν ότι οι ξένες ορδές ε, που δεν εισβάλλουν στη Βουλγαρία για να μείνουν, πολλοί θα ήθελαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να προχωρήσουν προς άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλήθεια πως οι συνθήκες υποδοχής στην Βουλγαρία, κύριε Κυρίλοφ, όσο και αν δεν σας αρέσει, έχουν φτάσει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο ε, που μόλις πρόσφατα άρχισε κάπως να βελτιώνεται και αυτό υπό τη διεθνή πίεση. Το ερώτημα για την Ευρώπη είναι το εξή και είναι κρίσιμο. Μιλάμε για την Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχουν 700.000 Σύριοι. 700.000 που φύγαν από τη χώρα τους. Εκτοπισμένοι εκατομμύρια μέσα στην ίδια τη χώρα ακόμα 750.000 στο Λίβανο που έφυγαν από την αιστεία του πολέμου και η Βουλγαρία τα ακούει γιατί δεν μπορεί να χειριστεί με λογικό τρόπο κάποιες χιλιάδες προσφύγων ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να υποδεχτούν λέει 50, άντε 500, άντε 1000 τι θα κάναμε αν έρχονταν 100.000 άνθρωποι ή 200.000 άνθρωποι Μα επιτέλους θα έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα έχει στόχο ε, ε, να υποδεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να τεθούν σε φυγή ή ακόμα μια φορά το Συμβούλιο κατά την ε, προσφυλή του συνήθεια θα αναβάλει το θέμα. Δεν πρόκειται αυτό να λύσει το πρόβλημα εάν προκύψει επίγουσα ανάγκη για τις μεταναστευτικές ροές. Σας ευχαριστώ κύριο Σκάλφιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα στη Βουλγαρία έχουμε 11.600 πρόσφυγες και η μισή είναι από τη Συρία. Η ροή των προσφύγων ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι και έχει συνεχιστεί και μέχρι τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Το Νοέμβριο 332 μπήκαν στη χώρα μας. 662 το Σεπτέμβριο. Η κρίση για την οποία λοιπόν συζητάμε είναι μια κρίση κάποιων μηνών. Ο κύριος Έγγελ είπε πώς τελείωσε. Δεν καταλαβαίνω για ποια κρίση μιλάει. Ανησυχώ για τα όσα μας είπε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέτρα τα οποία θα λάβει είναι μερικά και δεν είναι ορθά. Η Βουλγαρία χρειάζεται ένα μηχανισμό ε, επιπλέον που θα μας οδηγήσει σε συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία και θα πρέπει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να αναλάβουν και ένα μέρος αυτών των προσφύγων. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε τη Βουλγαρία για να υποδεχθεί αυτούς τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, δέκα φορές παραπάνω από τον αριθμό τον οποίο θα μπορούσαμε εμείς να υποδεχθούμε. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί πως είναι αμερόληπτη, τότε να αναλύσει την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Βουλγαρία. Η κυρία Γκαμπριέλε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διαπίστωσε πως έχουν ληφθεί κάποια μέτρα υπέρ των προσφύγων. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την τόλμη και το θάρρος ε, για να δηλώσουμε ξεκάθαρα πως η Βουλγαρία δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει αυτή την πρόκληση. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ξενοφοβικά φαινόμενα τα οποία έχουμε στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε στρατηγική για το μέλλον και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ξέρετε πως λήγουν τέλη Απριλίου. Το πρόβλημα λοιπόν θα ξεσπάσει και πάλι και ξέρετε τι συμβαίνει με εφήβους, με παιδιά, που ταξιδεύουν προς τη χώρα μας. Δεν θέλω να κάνω ερωτήματα χωρίς να δίνω απαντήσεις, αλλά πώς θα εντάξουμε τα άτομα αυτά στην κοινωνία μας αργότερα. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινότητες, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, στην επιμόρφωση των αστυνομικών και των συνοριοφυλάκων για να ξέρουν πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Συνεργασία λοιπόν με την Τουρκία για παράδειγμα και με ε, τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί από κοινού το πρόβλημα. Είναι πολλά τα μέτρα που χρειαζόμαστε. Κύριε Φαγιόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία με τους πρόσφυγες είναι πραγματικά τραγικά. Πρόκειται για τραγωδίες οι οποίες εκτελήσονται στα εξωτερικά σύνορα της Βουλγαρίας και αυτές οι τραγωδίες δοκιμάζουν την αλληλεγγύη μα Θα πρέπει να εισακούσουμε αυτές τις εκκλήσεις για βοήθεια και για αλληλεγγύη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να διωχθούν εκτός των συνόρων. Αυτή η απόφαση της Βουλγαρίας να υψώσει έναν έστω και προσωρινό φράχτη είναι πραγματικά κάτι αυτό που θέλουμε, να υψώνουμε τείχους και φράχτες στην Ευρώπη, θα πρέπει να γίνονται σε αυτά τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτό υπάρχουν μεταναστευτικές ροές και πιέσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε οι μηχανισμοί ελληνικής είτε άλλα μέσα για να διασφαλιστεί η βοήθεια προς τους ανθρώπους αυτούς, προς τις ομάδες αυτές που είναι ιδιαίτερω ευάλωτες, που μπορούν πραγματικά να έχουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα. Ο κύριος Δίας Νταμέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων άρθρου 33 και να ξεκινήσουμε επίσης το σχέδιο δράσης, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι επίγουσα, όχι, είναι έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ξεφύγει πια από το επίπεδο της ε, επίγουσας ε, ανάγκης και πρέπει να σας πω πως χρειαζόμαστε να δείξουμε αλληλεγγύη Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τρία βασικά στοιχεία. Στέγη, περίθαλψη και τροφή. Αυτά θα καλύψουν τις επίγουσες ανάγκες μας. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να συζητάμε ούτε το άσυλο ούτε τον έλεγχο των συνόρων. Γιατί τι μου λέει η δική μου εμπειρία από τέτοιου είδου πρόσφατου πολέμου πολέμους που έγιναν κοντά στην Ευρώπη. Δεν θέλουν οι Σύριοι να μείνουν στι χώρε μα. Θέλουν να σώσουν τη ζωή του και να γυρίσουν στη χώρα του. Άρα λοιπόν είναι απολύτω απαραίτητο να συνεργαστούμε, να δείξουμε αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μόνοι δεν θα τα καταφέρουν. Okay. Um, Τώρα θα πούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω διάφορους ομιλητές, όλοι είναι από τη Βουλγαρία και ο κύριος Κάζακ, ο κύριος θα έχει πρώτος το λόγο. Ήθελα να σας πω Αξιότιμοι συνάδελφοι, πως η κατάσταση στη Βουλγαρία μπορεί και να χειροτερεύσει. Και με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, συνεχίστε, είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό με τη Γερμανία. Θα ήθελα να σας πω πως η κατάσταση ενδέχεται να χειροτερεύσει, γιατί αν δεν βοηθήσουμε τις ΜΚΟ και αν δεν μας βοηθήσει ο ιδιωτικός κλάδος, δεν θα τα καταφέρουμε. Η Βουλγαρία, οι θεσμοί της δεν ήταν προετοιμασμένοι για τέτοια εμβέλεια κρίση. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η, βαρύνη, η ευθύνη βαρύνει την κυβέρνηση τούτη και την προηγούμενη, αλλά αυτά τα άτομα, αυτές οι οργανώσεις οι οποίοι μας βοήθησαν αυθόρμητα, οργανώθηκαν σωστά και κατάφεραν να μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι τόσο καλά οργανωμένοι που πολλές φορές ε, οι διεθνείς οργανισμοί μας λένε πως ε, τα πάμε υπερβολικά καλά. Λοιπόν, μας είπατε πως είναι αδύναμοι οι θεσμοί μας Κύρια Μάλστρομ, σας παρακαλώ, μην χαλαρώσετε τον έλεγχο που κάνετε στη βουλγαρική κυβέρνηση. Η Βουλγαρία δεν είναι έτοιμη και δεν έχει εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτό αληθεύει. Όμως θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη θέληση, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα εξαφανιστεί χωρίς συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορούμε να αφούμε ε, ε πως απλώς είμαστε αισιόδοξοι, πως κάποια στιγμή θα λύσει η σύραξη, θα λήξει η σύραξη στην ε, Συρία. Το πρόβλημα θα παραμείνει στην επικαιρότητα και πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Επίτροπε, η Ένωση καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ένα ψήφισμα για τη Συρία μετά από την ε, Λαμπετούζα. Ξέρετε, τις ημερομηνίε όπου συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα. Φυσικά το, η Βουλγαρία έχει πρόβλημα, δεν είναι άμεσο γείτονα τη Συρία. Οι πρόσφυγε πρέπει να διασχίσουν ολόκληρη την Τουρκία για να φτάσουν στη Βουλγαρία. Το πρόβλημα είναι ότι 50% των ανθρώπων αυτών είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Μετανάστες που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική και άλλες χώρες και αυτό αποτελεί πηγή κινδύνου για τη Βουλγαρία και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βία περιστατικά όπου εμπλέκονταν μετανάστες είναι γεγονότα. Ε, επίσης υπάρχει τάση ε, ξενόφοβων ε, εκδηλώσεων ξενόφοβων φαινομένων και η Βουλγαρία δεν μπορεί αυτά τα προβλήματα να τα λύσει μόνη του. Ε, μπορεί να είναι αλήθεια ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν και στατιστικές. Από τον Αύγουστο η Βουλγαρία εγγυάται τι συνθήκε για να υποδεχτεί χιλιάδες προσφύγων και συνεχίζει να το κάνει. Μένβα. Κυρία Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου βασίζεται στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Η Βουλγαρία πληρεί αυτές τις δύο, τους δύο όρους. Η χώρα μας δέχεται μεγάλες πιέσεις, αλλά τα προβλήματα των πρώτων ημερών έχουν ξεπεραστεί. Εμείς σεβόμαστε τον κανονισμό του Δουβλίνου και εργαζόμαστε για τη διαχείριση της χρήσης μαζί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, μέσα σε πλήρη διαφάνεια. Μάλιστα, κύριε Επίτροπε, πολλές προσπάθειες θα πρέπει ακόμα να γίνουν για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, αλλά και για να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική ε, διαδικασία για την εξέταση των ε, Όμω η Βουλγαρία μέχρι στιγμή δεν βασιζόταν παρά μόνο στα δικά τη μέσα. Τον Ιανουάριο λάβαμε την πρώτη οικονομική βοήθεια από την Ένωση και χάρη στην αλληλεγγύη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη βοήθεια των βουλγαρικών ε, διοικητικών μηχανισμών είμαι βέβαιη πως και χωρίς το 33 θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ κύριος Κυρίλοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψατε μου να υπογραμμίσω ότι με ευχάριστα από τα όσα είπαν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση η συμπάθεια αυτή που εκφράστηκε ακόμα και μέσω επικρίσεων γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να λύσουμε προβλήματα όχι μόνο σημερινά αυτά που είναι δηλαδή ε, τα σημερινά και επίκαιρα αλλά και τα μελλοντικά προβλήματα διότι τα βουλγαρικά σύνορα είναι σύνορα εξωτερικά της Ένωσης και εκτείνονται σε 200 χιλιόμετρα. Και πρέπει να λυθούν πολλοί άριθμα προβλήματα. Ευχαριστώ την Επίτροπο Μάρστρομ που τα υπογράμμισε όλα αυτά. Υπογράμμισε επίσης ε, την απαραίτητη ενεργοποίηση του μηχανισμού αλληλεγγύης, διότι εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλα αυτά αν κάθε κράτος μέλος δεν αντιδρά αντίστοιχα ανάλογα με ε, τον πληθυσμό του και το ΑΕΠ του και ευχαριστώ τον Έλληνα Υπουργό διότι είναι μια εμπειρία πολύ χρήσιμη ε, για τη Βουλγαρία και γνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από όλες τις μεσογειακές χώρες και πόσο οι πληθυσμοί μας είναι ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που λαμβάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι η αλληλεγγύη για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριο Κάζακ. Καζάκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κρίση με τους πρόσφυγες στη Βουλγαρία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013. Εμείς εγκρίναμε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης και το 85% των μέτρων από το σχέδιο αυτό έχουν εκτελεστεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Ο αριθμός των προσφύγων που έχουν περάσει λαθρέα τα βουλγαρικά σύνορα ε, μειώνεται και μπορούμε να πούμε πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μαζικές ροές πια. Ο αριθμός των ατόμων που ε, ζητούν άσυλο σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί πολύ. Η κυβέρνησή μας λοιπόν αντέδρασε και αντέδρασε με το σωστό τρόπο. Δεν είχαμε ούτε επιδημίες, ούτε μολυσματικές ασθένειες, ούτε ε, ανθρώπους να ζουν σε σκηνές μες στο χειμώνα. Ξέρετε πόσο ο αριθμός των προσφύγων το 2013 ε, αυξήθηκε ραγδαία η Βουλγαρία και αυτό αποδεικνύει ε, πως, ε, κυρία Επίτροπε, μπορεί μόνη της και χωρίς το άρθρο 33 να πορευτεί η χώρα μας. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγα πρόεδρε τη μετάφραση, Λοιπόν, που καθυστερήσα. Όντω, ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε αποστολή και εμεί ε, έχουμε μεταβεί συχνά στη Βουλγαρία. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στη Βουλγαρία σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφτασαν στη χώρα πάρα πολλά άτομα και δεν ε, ήταν προετοιμασμένη η χώρα. 11.000 άτομα έφτασαν πέρσι. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι για μια χώρα που δεν έχει την υποδομή να τους υποδοχτεί. Είναι πολλοί λοιπόν αυτοί στη Βουλγαρία και φυσικά είναι ανάλογοι αυτοί, αυτός ο αριθμός ανθρώπων που καταφτάνουν κάθε εβδομάδα με αυτού που καταφθάνουν κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα, στη Γερμανία και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν πάρα πολύ σημαντικά μέτρα. Είναι ανησυχητική η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλε ευρωπαϊκές υπηρεσίε, τα κράτη-μέλη, διεθνεί οργανώσεις, παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Είναι σαφές ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί η πίεση στα εξωτερικά σύνορα, γιατί δεν θα επιληθεί η κατάσταση στη Συρία αύριο. Και να πω ότι το ίμιση ε, από τα άτομα αυτά που έχουν καταφτάσει είναι από τη Συρία. Οι υπόλοιποι είναι από Αφγανιστάν, από το Πακιστάν και από άλλες χώρες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί, πολλές χώρες που υπόκειται πιέσει στην γειτονιά μας. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ακόμα σε ό,τι αφορά ε, τις όρους ε, υποδοχής, ε, τα καταλήματα, ε, ένταξη για όσους έχουν λάβει το δικαίωμα να μείνουν, που θα μείνουν και κατά πάσα πιθανότητα για πολύ καιρό στη Βουλγαρία και σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν τα σύνορα, που και εκεί γίνεται δουλειά. Αλλά όπως είπε η κυρία Γκυγιόμ, θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στον κόσμο να προσέρχεται στα σύνορα και να ζητά άσυλο. Έχουμε ακούσει και σε ό,τι αφορά τι βουλγαρικέ αρχέ, ότι οι οι αποθήσει είναι παράνομε. Θα πρέπει λοιπόν να διεξαχθεί ένα τέτοιο διάλογο. Είναι λοιπόν τρομακτικό αυτό ο πόλεμο πολύ κοντά στην Ευρώπη, στη Συρία. Οι όμορε χώρε ε, τη Συρία έχουν και φέρουν τεράστιε ευθύνε. Περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγε ε, έχουν υποδεχτεί έχουν ανοίξει τα σύνορά τους. Πολύ μικρός είναι ο αριθμός των προσφύγων αυτών που έχουν έρθει στην Ευρώπη. Αν, έχουν, αν συνέβαλαν και 28 χώρες θα μπορούσαμε να υποταχθούμε πιο πολλά άτομα. Η πιο άμεση βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στη Συρία είναι να ανοίξουμε τα σύνορά μας για τέτοια πρόσβαση στις χώρες μας με νόμιμο και ασφαλή τρόπο προκειμένου ο κόσμος αυτός να μην ε, προσφεύγει σε επικίνδυνες μεθόδους για να διασχίσει τη Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω λοιπόν την έκκλησή μου προς όλα τα κράτη-μέλη και προς τα 28 κράτη-μέλη να υποδεχτούν τέτοιους πρόσφυγες από την περιοχή. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να συνδράμουμε τους πιο ευάλωτους ε, σε αυτή την ε, εποχή, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν παράλληλα να επιδείξουμε και αλληλεγγύη με την Βουλγαρία για να βοηθήσουμε την Βουλγαρία να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος ο κ. Μανιζέλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιλαμβάνονται την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. είμαστε χώρα γειτονική προς τη βουλγαρία χώρα με τεράστια ακτογραμμή υφιστάμεθα και εμείς όπως και όλες οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες πολύ μεγάλες πιέσεις καθημερινές πιέσεις στα θαλάσσια σύνορά μας και στα χερσαία σύνορά μας. η βουλγαρία πράγματι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οξύ πρόβλημα εντοπισμένο στα χερσαία σύνορά της το πόλεμο αυτό μας οδηγεί στο να κατανοήσουμε πόσο κρίσιμο είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συνεργασία ευρωπαϊκής ένωσης και τουρκίας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η συμφωνία επανεισδοχής που υπεγράφει πριν από λίγες εβδομάδες ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ένωση και την τουρκία. τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί στην πράξη το αξίωμα το δόγμα της δίκαιης και αναλογικής κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη μέλη. αυτό είναι συνυφασμένο με την αλληλεγγύη ως βασική αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. βέβαια στις συζητήσεις στο επίπεδο του συμβουλίου η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζεται αφενός μεν ως ένα οξύ ανθρωπιστικό πρόβλημα ως διαχείριση μιας διαρκούς οξείας ανθρωπιστικής κρίσης αντιμετωπίζεται και ως πρόβλημα ασφάλειας γιατί πίσω από την ανθρωπιστική πίεση από αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη βοήθειας από αυτούς που ζητούν άσυλο από αυτούς που μπορούν να χαρακτηριστούν πράγματι πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που θέτουν ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι επίσης πολύ σημαντικό να τονίσω ότι η αντιμετώπιση του θέματος αυτού κινείται σε δύο επίπεδα παράλληλα. το πρώτο επίπεδο είναι τα άμεσα μέτρα η αντιμετώπιση της κατάστασης επί του πεδίου τώρα που υπάρχει το πρόβλημα γιατί το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να περιμένει και εκεί χρειάζονται πρακτικές μορφές αλληλεγγύης και στήριξης χωρών όπως η βουλγαρία. υπάρχει και το άλλο επίπεδο του συνολικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. η προεδρία του εξαμήνου αυτού που έχει ήδη συνεργαστεί και με την επόμενη προεδρία της ιταλίας έχει θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα αυτό γιατί ε, πρέπει πράγματι η ευρώπη να δείξει την ικανότητά της να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ζητήματα αυτά. θυμίζω ότι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του οκτωβρίου έγινε μια πρώτη συζήτηση σε βάθος για το πρόβλημα αυτό υπό την πίεση της ανθρωπιστικής κρίσης του δράματος μάλλον της λαμπεντούζα. στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του δεκεμβρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ομάδας δράσης για τη μεσόγειο. πριν από λίγες μέρες στην αθήνα στις 24 και 25 ιανουαρίου οργανώθηκε η άτυπη υπουργική σύνοδος δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συμμετοχή της κυρίας Μάλστρομ και εκεί έγινε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης σε συνέχεια και των συμπερασμάτων της ομάδας δράσης για τη μεσόγειο. έχουμε μια καλή αξιόπιστη βάση προκειμένου να διαμορφώσουμε στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο μετά τη στοκχόλμη. βεβαίως περιμένουμε τη σχετική ανακοίνωση της επιτροπής ελπίζουμε το μάρτιο έτσι ώστε το αργότερο στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του ιουνίου να υιοθετήσουμε στρατηγικές κατευθύνσεις για το ζήτημα αυτό η καθημερινή διαχείριση του προβλήματος στη βουλγαρία όπως και στην ελλάδα στην ιταλία στη μάλτα δεν μπορεί φυσικά να περιμένει ούτε τον μάρτιο ούτε τον ιούνιο είναι κάτι που διεξάγεται καθημερινά υπό συνθήκες πίεσης συχνά δραματικές. εκεί νομίζω ότι κατανοήσαμε και από τις παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα στη συζήτηση τι πρέπει να γίνει. η επιτροπή έδωσε τη δική της απάντηση. θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα μεταφέρω στο συμβούλιο τις παρατηρήσεις και την αγωνία που εκφράστηκε εδώ από όλους τους ομιλητές όχι μόνο όσους ζουν ως βούλγαροι πολίτες το πρόβλημα αλλά γενικότερα από όλο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γιατί εδώ δοκιμάζεται η κοινή ευρωπαϊκή συνείδησή μας. ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Όλους τους ομιλητές, έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και τώρα περνάμε στη συζήτηση για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Όπου πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Βενιζέλος.